εννοείται ότι είναι προτεραιότητα και τη Προέδρου Φοντερ Λάιεν και μάλιστα σημειώσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Αντιπρόεδρος Γιώροβα θα είναι αρμόδια για το συντονισμό του σχεδίου δράση για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλειών. Κάτι τέτοιο ε, ε, προϋποθέτει την εστίαση στην ενίσχυση τη ανθεκτικότητα και στην προάσπιση των ε, θεμελιωδών ελευθεριών. Η αντιμετώπιση βρυδικών ε, απειλών χρήζει οριζόντιας προσέγγισης και μεθόδων και φυσικά στενή συνεργασία και συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στα κοινοτικά θεσμικά όργανα αλλά και στα κράτη-μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των κρατών μελών να προλάβει, εντοπίσει και να ανταποκριθεί, να καταπολεμήσει υβριδικέ απειλέ. Η προστασία τη δημοκρατία και των εκλογών προποθέτει συντονισμένε δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών, αλλά και ε, ανάμειξη τη κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία. Η απάντησή μα θα πρέπει να είναι συνολική και να, έχει και εσωτερική, να λαμβάνει υπόψη και την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της απειλής. Πολλά έχουν γίνει ήδη από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αλλά και από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Και θα αναφερθώ σε κάποια ορόσημα που είχαμε στην προσπάθεια αυτή, όπως τις τακτικές απαφές στο δίκτυο ε, εκλογών, ε, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ενίσχυση στρατηγικής επικοινωνίας, διευκόλυνση των δικτύων ανεξάρτητων ε, φορέων ελέγχου της εγκυρότητας, ε, εξτρατείες ευαισθητοποίησης, ε, ψηφιακός γραμματισμός και καλύτερο συντονισμό των πρακτικών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά χρειάζονται και περαιτέρω θεσμικοί μηχανισμοί και εργαλεία για να υλοποιήσουμε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και κυρίως ε, τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Αντιμετώπιση βρετικών Απειλών του Ελσίνκη συμμετέχει στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα αυτό. Επίσης, ε, οι στρατηγικές παραπληροφόρησης ξένων παραγόντων λαμβάνουν χώρα και εκτός των σύνορων μας, οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε με εταίρους μας της ε, νότιας και ανατολικής γειτονίας, αλλά και των εταίρους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου μήνα αναφέρεται ε, η παραπληροφόρηση, ο σωστό έλεγχος της ε, χρηματοδότησης ε, των πολιτικών μηνυμάτων, ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία των συμπερασμάτων. Θα πρέπει να δράσουμε από κοινού με συγκροτημένο και συντονισμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τις απειλέ. Η διαφύλαξη των εκλογών βρίσκεται στο επίκεντρο της προάσπισης των ευρωπαϊκών μας αξιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Κομισιόν και σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Τον λόγο κύριε Γιώργα. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρέμβω για αυτό το ζήτημα της παρέμβασης άλλων χωρών στις δημοκρατίες μας και στις εκλογές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται, έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τους πολλούς και διάφορους κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη διαφάνειας, την παραπληροφόρηση, και άλλες μορφές χειραγώγησης εκλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών. Και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια στην επόμενη θητεία. Και βεβαίως, όπως είπε και η Προεδρία, θα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες ε, του χαρτοφυλακίου μου και ευχαριστώ για την στήριξη. Οι δίκες ε, και ελεύθερες εκλογές είναι ένα θέμα ευθύνης των κρατών μελών, η διεξαγωγή τους. Βεβαίω χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, διότι η διασυνοριακή διάσταση ε, στην χειραγώγηση τη δημοκρατία ε, και η σημασία του να ενώσουμε τι δυνάμει μα για να αντιμετωπίσουμε τι απειλέ ε, είναι κάτι το οποίο είναι πλέον προφανέ. Κάτι που επηρεάζει ένα κράτο μέλο, Το επηρεάζει όλα. Επηρεάζει, έχει ένα αντίκτυπο στο σύνολο τη Ένωση. Οι απειλέ αυτέ είναι περίπλοκε και εξελίσσονται συνεχώ. Παραδείγματο χάρη, οι εξωτερικοί παράγοντες πολύ συχνά χρησιμοποιούν εσωτερικούς εκπροσώπους. Υπάρχουν και εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες που δίνουν ε, δυνατότητες για νέες μορφές και στρατηγικές παρέμβασης. Στα πλαίσια των εκλογών του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις ένα πακέτο μέτρων για τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Ευρώπη, κώδικας των ε, πρακτικών που δημιουργήθηκε σε πέτο Facebook, ε, Twitter ε, και άλλων πλατφόρμων. Επίσης, έχει σημειωθεί πρόοδος ό,τι αφορά τη δράση κατά της παραπληροφόρησης. Και βεβαίως σε αυτό επάνω θα βασιστούμε στην επόμενη θητεία. Προσπαθούμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση και μια μόνιμη μορφή αντίστασης για να μπορεί να είναι ανθεκτική η δημοκρατία μας απέναντι σε απειλές οι οποίες ε, εξελίσσονται ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη χειραγώγηση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές λοιπόν χρειάζεται μια συντονισμένη και σφαιρική προσέγγιση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα, κοινοβούλια, ρυθμιστικές αρχές, αρχές εφαρμογής του νόμου, δημοσιογράφοι, πολιτικά κόμματα, ερευνητές, εκπαιδευτέ κοινωνία των πολιτών γενικότερα, καθώς και η βιομηχανία βέβαιως και, βεβαίως και οι επιγραμμικές πλατφόρμες. Κάποιες αναφέρονται και συμμετέχουν ήδη, αλλά πρέπει να έρθουν και άλλες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή. Και βεβαίως χρειαζόμαστε και τους πολίτες. Πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να γίνουν πιο ανθεκτικοί απέναντι στις νέες απειλές. Ορισμένες φορές λέω ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση για την αλήθεια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο καθήκον που μας περιμένει. Θα πρέπει να εντοπίζουμε, να αναλύουμε, ε, να καταδεικνύουμε αυτές, αυτή την παραπληροφόρηση στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιες και αν είναι οι τακτικές που χρησιμοποιούνται. Και αυτό πάει χέρι-χέρι με μια ευρύτερη προσπάθεια για την παρακολούθηση της κυβερνοασφάλειας και την ανθεκτικότητα κατά των υβριδικών απειλών. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, Υπάρχει μια πολύ, ένα πολύ καλό δίκτυο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τις εκλογές που συνεργάζεται σήμερα για πέμπτη φορά και που θα εξετάσει τις μελλοντικέ του δράσεις απέναντι ε, για την προάσπιση μάλλον των εκλογών είναι ένα πολύ σημαντικό νέο εργαλείο στην εργαλειοθήκη μα. Θα πρέπει να αυξηθεί επίση η συνεργασία μεταξύ εθνικών οργάνων τη Ένωση και κρατών μελών μέσω αυτού του δικτύου. Να υπάρχει ένα συστημάκι τη προειδοποίηση που θα μα βοηθήσει ε, με τη συμμετοχή ε, μιας μεγάλης κοινότητας ε, εμπειρογνωμών. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με εταίρους όπως το G7, όπως το ΝΑΤΟ, διότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσω μιας συντονισμένης απάντησης απέναντι στις, τα επεισόδια παραπληροφόρησης, να αυξηθεί γενικότερα η ευαισθητοποίηση του κοινού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθειά μας για να διευκολύνουμε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης κοινότητας ανθρώπων που ελέγχουν τα γεγονότα, ε, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ε, σε ό,τι αφορά αυτά που συμβαίνουν στα κοινωνικά, δίκτυα, στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Ο κώδικας ορθών πρακτικών ε, αυτή τη στιγμή αξιολογείται μετά από μια πρώτη ε, περίοδο λειτουργία, εάν δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, η Κομισιόν ενδεχομένω να προτείνει περαιτέρω μέτρα και ρυθμιστική φύσεω. Θα πρέπει επίση να ενισχύσουμε ε, τον αλφαβητισμό ε, όσων ε, παρακολουθούν τα μίντια. Θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να συμμετέχει κάποιο στι δημοκρατικέ διαδικασίε σωστά ενημερωμένο. Η νέα πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε νέο, μια νέα νομοθεσία για τι ψηφιακέ υπηρεσίε που θα αυξήσει του κανόνε ασφαλεία και αξιοπιστία των πλατφόρμων αυτών και την, που, που πολλούν και προϊόντα και υπηρεσίε. Πρέπει να έχουμε επίση μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουν να βοηθήσουν για να εξασφαλίσουμε ένα ε, ασφαλές μέλλον σε ψηφιακό επίπεδο για την Ευρώπη. κυρία Φόντερ Λάιεν ε, και εγώ θα εργαστούμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχέδιου Δράση για τη Δημοκρατία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των παρεμβάσεων στι εκλογέ μα. Πάντα βέβαια ε, θα έχουμε κατά νου και την προστασία του δικαιώματο έκφραση. Θα εξετάσω τι ενδεχόμενε νομοθετικέ προτάσει έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σαφέστερου κανόνε για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και μεγαλύτερη διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ διαφημίσει δεν πρέπει ποτέ όμως να χάνεται το σημείο ισορροπίας. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις, ευρωπαϊ... τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες μας, οπότε ο σεβασμός της ελευθερίας έκφρασης και των θεμελιών δικαιωμάτων και των αξιών μας πρέπει να είναι κάτι που θα μας απασχολεί διαρκώς. Ευχαριστώ. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin Nun nächstes für die EVP-Fraktion. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Ρανζέλ για το ΕΛΚ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην εκπρόσωπο της Φιλανδικής Προεδρίας ευχαριστώ να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο Βέρα Γιώροβα για την εκλογή της, να της ευχηθώ καλή τύχη και να της πω ότι γνωρίζω απόλυτα ότι είναι απόλυτα προσιλωμένη ε, στο έργο της και στο καθήκον της. Ε, το χαρτοφυλάκιο της είναι περίπλοκο, αλλά πραγματικά ξέρω ότι είστε ενθουσιώδεις και προσιλωμένοι. Σας εύχομαι καλή τύχη, καλή επιτυχία και μπορείτε να υπολογίζετε στην ε, συνεργασία της ομάδας αλλά και του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε αμέριστα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Η απόπειρα παρέμβασης είτε από εξωτερικές δυνάμεις, από ξένες δυνάμεις, είτε από κάποια συνενοχή μεταξύ εσωτερικών δυνάμεων, αυτή η παρέμβαση είναι αναμφίβολα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η παραπληροφόρηση δεν είναι κάτι καινούριο στην ιστορία, δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά έχουμε λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων τεράστια ε, απήχηση της παραπληροφόρησης σε όλη την κοινωνία και μεγάλη επιρροή της. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι πρόσφατα οι τσεχικές μυστικές υπηρεσίες ε, πέσαν την προσοχή μας ε, στο πρόβλημα της κινέζικης και ρωσικής παρέμβασης σε εκλογικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε ότι και στο Brexit είχαμε τέτοια παρέμβαση. Γνωρίζουμε ότι και στην Καταλανία ένα σημαντικό τμήμα των ε, των διαδικασιών επηρεάστηκε από πράκτορες ε, Ρώσους. Επίσης, ε, γνωρίζουμε ότι έχουμε μερικές φορές και εσωτερική δυναμική και διαστάσεις που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από εξωτερικές δυνάμεις για να εντείνουν την πόλωση και την ρήξη των κοινωνιών μας. Οπότε είναι αποφασιστική σημασία και θεμελιώδου σημασία να μεριμνήσουμε κυρίως για την σωστή ενημέρωση των πολιτών, σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών και να αναπτύξουν αξιολογική κρίση ώστε να μπορούν να διαχωρίζουν ε, την ε, σωστή πληροφορία από την ανακριβή και την παραπληροφόρηση. Επίσης, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι επιστήμονες, οι πανεπιστημιακοί, οι ακαδημαϊκοί και οι δημοσιογράφοι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να αναπτύξουν μια ε, σωστή επαλήθευση των πληροφοριών για να μεταδίδονται σωστά οι πληροφορίες και η ενημέρωση στην κοινωνία. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, με τις χώρες που έχουν εντοπίσει τέτοιε παρεμβολές και παρεμβάσεις και να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε και εσωτερικές παρεμβάσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την περίπτωση της Μάλτας. Εκεί είχαμε την δολοφονία της δημοσιογράφου Δάφνε Καλίσια. Αυτό ήταν πραγματικά εξωφρενικό, τρομακτικό και δείχνει σε τι κίνδυνο βρίσκεται η ελεύθερη πληροφόρηση. Ε, μερικές φορές ε, υφίστε και προσωπικούς κινδύνους και ψηφιακούς και σωματικούς. για τους σοσιαλδημοκράτες, κυρία Κάτι πήρε για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, συγχαρητήρια και από εμάς. Οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι η καρδιά της δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και της Ένωσης, αλλά οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές δεν είναι κάτι το δεδομένο. Η παρέμβαση στις εκλογές ε, αμφισβητεί τα θεμέλια του δημοκρατικού συστήματος και είναι ένας κίνδυνος που αυξάνεται καθημερινά και πρέπει να κάνουμε κάτι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πολιτικές ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν αυτήν την υβριδική επίθεση στην δημοκρατία. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτίθενται σε τεράστιες εκστρατείε παραπληροφόρησης λόγω της ξένης παρέμβασης. Οι κυβερνοεπιθέσει έχουν φτάσει πρωτοφανή επίπεδα και πλέον κινδυνεύουν οι στρατηγικέ υποδομέ και τα δεδομένα και οι εκλογικοί κανόνες ε, για την χρηματοδότηση κομμάτων από τρίτες χώρες παραβιάζονται. Όμως οι κυβερνήσεις της Ένωσης ακόμα δεν δρουν. Κάποιες κρύβουν την αλήθεια από το κοινό. Αυτό συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον παραδείγματος χάρη. Προσφάτως αρνήθηκε να δημοσιεύσει την έκθεση της Επιτροπής Μυστικών Υπηρεσιών για την παρέμβαση στις Βρετανικές εκλογές. Όμως δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Οι Ρώσοι είχαν χρηματοδοτήσει την Λίγκα του Σαλβίνη, το FPE, ε, το Front National, την εκστρατεία Λίβ στο Ηνωμένο Βασίλειο και διάφορες άλλες ύποπτες δραστηριότητες στη Γερμανία. Τον προηγούμενο μήνα, μετά από πρωτοβουλία της ομάδας μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έκανε ένα ψήφισμα όπως ζητήσαμε να αναλυφθεί η δράση και στο Κοινοβούλιο. Αντιλαμβανόμαστε την σημασία αυτού του ζητήματος και ζητάμε να συσταθεί μια ειδική επιτροπή για το θέμα αυτό για να δει το ζήτημα συνολικά. Αλλά η πρόταση δεν πέρασε λόγω της αντίδρασης 52 συναδέλφων του Ρινιού. Και απορώ γιατί οι συνάδελφοί μας από το Ρινιού και πιο συγκεκριμένα οι φιλελεύθεροι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν δέχτηκαν να μπει το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη και καταψήφισαν την σύσταση της ειδική Επιτροπής. Όμως, καμιά φορά βεβαίως τα πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους. Ας συνεργαστούμε λοιπόν έτσι ώστε να φροντίσουμε ότι θα πάρουμε το ζήτημα αυτό στα σοβαρά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντουιράν για την ομάδα, η κυρία Ντουιράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω για την επανακλογή σας σήμερα το πρωί και θα ήθελα να πω προσωπικά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβρίσκω εδώ για τα ζητήματα που μας είχαν ήδη απασχολήσει στα πλαίσια της προηγούμενης θητείας και πιο συγκεκριμένα για το θέμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η ιστορία μας πάντα προσπαθεί να βρει το σημείο ισορροπία, το οποίο είναι περίπλοκο. Η κυρία Φοντελάιν αναφέρθηκε στο πόσο έθραυτε είναι οι δημοκρατίε μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ επειδή αναζητούμε ιστορικά αφενό την υπεράσπιση τη ελευθερία, των ελευθεριών, του δικαιώματο έκφραση, τη ελεύθερη σκέψη και αφετέρου το σεβασμό των κανόνων, του δικαίου που, ισχύουν για όλους, για να μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί στην ίδια κοινωνία εμείς μπορέσαμε να, ε, να εφεύρουμε ε, το, την τυπογραφία. Και χάρη στην τυπογραφία βελτιώθηκε η γνώση ε, των συμπολιτών μας. Περασπιστήκαμε την ελευθερία σκέψης, την ελευθερία του τύπου και μπορέσαμε να βρούμε και το σωστό σημείο ισορροπίας. Το γνωρίζετε πολύ καλά κυρία Πρόεδρε, διότι προέρχεστε από μια χώρα που όπου δεν υπήρχε πάντα ελευθερία σκέψης και ελευθερία έκφρασης. Μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε αυτό το σημείο ισορροπίας μέσω της αρχής της ευθύνη όσων διαδίδουν πληροφορίες και μέσω κανόνων που έχουμε επιβάλει στον τύπο και στο τι ε, μεταδίδει, τι διαδίδει. Δεν μπορούμε ε, να ε, διαδίδουμε τα πάντα. Και όταν έρχεται το ίντερνετ και αντικαθιστά τον τύπο και πάει πολύ πιο γρήγορα και μας εξηγεί ότι πρέπει να του δώσουμε πλήρη ελευθερία ότι δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε, ότι πρέπει να αυτορυθμίζεται το διαδίκτυο. Ε, λοιπόν, εγώ κυρία Αντιπρόεδρε λέω ότι εδώ πραγματικά πλήττεται η ουσία της αξίας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή το σημείο ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας και των κανόνων. Και τελειώνοντας να πω ότι δεν πρέπει το διαδίκτυο να γίνει ένας χώρος όπου δεν υπάρχει δίκαιο, ε, ας μην γίνουν τα, ε, τα κοινωνικά δίκτυα δικτύωσης ένας χώρος ελευθερίας χωρίς κανέναν έλεγχο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο συνάδελφος Λαγκοντίνσκι από τους Πράσινους. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και από τους Πράσινους στην κυρία Αντιπρόεδρο για την εκλογή της. Σήμερα όμως μιλάμε για ένα άλλο θέμα. Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ε, καταστρέφει την οικονομία μας. Ε, αυτό ήταν ο τίτλος ενός email ο οποίος παρέλυσε το σύστημα email της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας μέσω ενός ε, ιού. Και ήταν κάτι το οποίο έστειλαν οι ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες. Το πιο απτό και προφανές παράδειγμα παρέμβασης ε, στα δημοκρατικά μας ε, θεσμικά όργανα. Πολλά όμως περνάνε χωρίς να τα προσέξουμε και είναι ανισχυτικά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα παρέμβαση και έχουμε μια πραγματική ιδεολογική αντιπαράθεση, έναν πόλεμο προπαγάνδα στον ψηφιακό τομέα μεταξύ, πρέπει να το πούμε, Ρωσίας, Κίνας και των φιλελεύθερων δημοκρατιών από την άλλη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα γερμανικά και στα αγγλικά, αλλά και στα ρωσικά. Η περίπτωση Λίζα στην ε, χώρα μου, όπου κινητοποιήθηκαν πάρα πολλοί ρωσόφωνοι μέσω ειδήσεων στην ε, ρωσική τηλεόραση, ε, οι οποίες ήταν τελικά ψευδείς ειδήσει. Αλλά και στα αγγλικά και στα γερμανικά γίνεται αυτή η προπαγάνδα. Όχι μόνο στο Russia Today, το Redfish, στο Facebook, ένα ριζοσπαστικό δεξιό ε, site το οποίο από τη μία μιλάει για την πολιτική του κλίματος και από την άλλη κάνει προπαγάνδα και τα όσα μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορία. Και τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων πρέπει να δούμε επίσης. Και βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε και τους συναδέλφους μας εδώ πέρα. Έχουμε κόμματα που περιφρονούν βαθιά την ε, δημοκρατία και την Ευρώπη και κάθονται εδώ μέσα. Και σήμερα ήδη υπήρχαν κάποιες ειδήσει για το ΑΕΦΔ. Κρίμα που δεν είναι εδώ. Γιώργ Μόιντεν, 59.000. Γιέντε Ράιλ, 45.000. Αυτές είναι οι δωρεές ε, που έγιναν ε, για αυτούς τους συναδέλφους που κάθονται εδώ ανάμεσά μας. Πρέπει λοιπόν να τους ρωτήσουμε από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Μας λέει το ΑΕΦΔ ότι πηγαίνει στην ρωσική πρεσβεία για συνομιλίες. Πολλά από αυτά τα λεφτά ήρθαν μέσω Ελβετίας ε, και θα ήταν ενδιαφέρον να λάβουμε κάποιες απαντήσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οι αντιευρωπαίοι, το θέμα είμαστε και εμείς. Και εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα αυτή και εδώ πέρα βεβαίως πρέπει να έχουμε μια ουσιακή κουλτούρα και μια ανθεκτικότητα των θεσμικών οργάνων μας και εδώ και απέναντι στους συναδέλφους που μας χρωστάνε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Για το ID, ο συναδελφός Μπαρντέλα για να μισή λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγγνώμη έτσι που θα ε, γύρισω την πλάτη στην παράνοια που έχει ε, επιβληθεί εδώ. μα έχει επιβληθεί το θέμα αυτό διότι θέλουμε να πούμε ότι ο, η Ρωσία του Βλαδίμιρ Πούτιν κρύβεται πίσω από τι επιτυχίε των ε, εθνικών κινημάτων ανά την Ευρώπη. Αν ο κ. Μακρόν, η κυρία Μέρκελ χάνουν στι εκλογέ, αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο επειδή υπάρχει χειραγώγηση από το εξωτερικό. Η, το εθνικός, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας ε, των συστημάτων πληροφορική είπαν ότι δεν υπήρξε καμία κυβερνοεπίθεση από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εκλογών στη Γαλλία. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει καμία ε, εκστρατεία παραπληροφόρησης από το εξωτερικό που να αφορά ευρωπαϊκές εκλογές. Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι ε, βρίσκουν εδώ συνωμοσίε ε, είναι αυτοί που συνωμοτούν και που φαντάζονται ότι υπάρχει κάποιο αόρατο ρωσικό χέρι. Είναι σαφή, σαφές ότι υπάρχουν συνωμοσίες, αλλά προέρχονται από αλλού. Ο πρώην πρόεδρος ε, των ΗΠΑ, ο κ. Ομπάμα, δεν παρενέβη ανοιχτά στις γαλλικές εκλογές που προστηρίζονται τον κ. Μακρόν ανάμεσα στους δύο γύρους. Η κ. Μάρκελ, Μέρκελ ε, το 2017 ε, δεν είχε πει ότι θα πρέπει το Front National να, να υποχωρήσει και τι δεν έγινε για να μπορέσουν οι Βρετανοί να μην ψηφίσουν Brexit στις στα και τι, και δεν έγινε για να αποφευθεί η εκλογή του Σαλβίνη στην Ιταλία. Ε, εδώ μιλάμε για κάποιες, αιτίε, κάποιες αιτίες οι οποίες είναι σκοτεινές, οι οποίες δεν είναι ορθολογικές και οι οποίες ουσιαστικά δεν υπάρχουν και δεν καταλαβαίνετε ουσιαστικά οι ευρωπαϊκοί λαοί τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για το ECR. Ο κύριος Λούντγκριν για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δημοκρατίες μας ε, ανησυχούν πολλούς. Ε, σκεφτόμαστε τις αμερικανικές εκλογές, η χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν, η Ρουσία, ε, που θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν. Στην Σουηδία βέβαια ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με την Κίνα που προσπάθησε προσφάτως να επηρεάσει έναν υπουργό και την κυβέρνηση για να μην βραβεύσουν ένα άτομο το οποίο δεν είναι αρεστό στο κινέζικο καθεστώς. Ε, βεβαίως ε, ε, βλέπουμε ότι η Κίνα προσπαθεί να επηρεάσει τους άλλους και την διεθνή κοινή γνώμη. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η προσπάθεια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προπαγάνδα για να επηρεάσει τις εκλογές, λέγοντας ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Μιλάνε συχνά για μια και ζωγραφίζουν μια εικόνα η οποία είναι πραγματικά αποκαλυπτική για καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πόσο φοβερό και τρομερό θα ήταν αυτό. Μια προπαγάνδα δηλαδή που βασίζεται στον τρόμο για να επηρεάσει τις εκλογές. Αλλά θα πρέπει πραγματικά ε, ψάχνουμε να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτών ε, των πραγμάτων. Όχι, αλλά από την άλλη δεν σεβόμαστε και τα αποτελέσματα των εκλογών εδώ πέρα και αναζητούμε μόνο τι κάνει η Κίνα και η Ρωσία. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΥΕ, κυρία Άντερσον, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ξένη παρέμβαση σε εκλογικέ διαδικασίε και να μην εγκαλούμε το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα που ποτέ δεν λογοδότησε όταν εισέπραξε μισό εκατομμύριο λίρες ερλίνες μαύρο χρήμα κατά τη διάρκεια ε, τη εξτρέα του Brexit. Μαύρο χρήμα που δόθηκε στον DUP μέσω κάποιου υποτιθέμενου διεθνούς επιχειρηματία. Τα χρήματα αυτά δεν τα ξόδεψαν στη Βόρεια Ιρλανδία. Αντίθετα, το DUP τα ξόδεψε σε μια χώρα που δεν κατέβαζε υποψηφίωση, στην Αγγλία, προκειμένου να παρακάμψει εκλογικό ε, νόμο στην Αγγλία. Δεν έγινε καμία έρευνα για το, την προέλευση των χρημάτων αυτών. Και μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit θεσπίστηκε νομοθεσία ώστε να βρεθεί στο απειρόβλητο το DUP και να μην χρειαστεί να κάνει δήλωση υπόθενε έσχεση. Και αυτό είναι το DUP το ίδιο που έκανε παρένεση σε ενωτικά πλήθη να ψηφίσουν ε, υπέρμαχους του Brexit από το DUP. Και μάλιστα ανήρτησαν εκφοβιστικά πόστερ κατά του υποψηφίου και ε, του Σιν Φέιν και ε, δήμαρχου του Μπέλφας, του Τζον Φουνικέιν, ο πατέρας του οποίου δολοφονήθηκε από Βρετανούς πράκτορες και ενωτικούς. Αν γινόταν οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το καταδικάζαμε. Κι όμως ε, η διχοτόμηση της Ιρλανδίας που έγινε από ένα μιαρό μικρό δογματικό κράτος με μια ε, πλειοψηφία των ενωτικών ε, με στόχο την οθεία εκλογών και για να παρεμποδίσει την δημοκρατική βούληση των ανθρώπων ένα κράτος με αποκλεισμούς που θα ζήλευε ακόμη και η Νότια Αφρική του Απαρτχάιτ. Ευτυχώς όμως αυτό το λεγόμενο πορτοκαλί κράτος με την γενή ε, πλειοψηφία των ενωτικών έχει φύγει και βοδεύουμε προς μια ενωμένη χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατική Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ Λέναρς. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Το θέμα εδώ πέρα δεν ε, αφορά μόνο τις ε, εκλογές και πριν από ένα μήνα και πριν από δύο μήνες τα ξαναείδαμε λόγω των εκλογών και το ξαναβλέπουμε σήμερα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και δεν έχει αναλυφθεί καμία δράση. Πέρασαν οι ευρωεκλογέ. Είδαμε διάφορε έρευνε, ε, από τι οποίε προκύπτει ότι σχεδόν η μισή Ευρωπαίοι κατά τη ε, διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έπεσαν θύματα ε, παραπληροφόρησης από ρωσικά τρόλ. Ε, βλέπουμε σελίδες ε, ολόκληρες οι οποίες ε, εξαφανίζονται από το Facebook βεβαίως, αλλά πρώτα τις έχουν δει εκατοντάδες εκατομμύρια φορές οι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν και την Task Force Στρατηγικών Επικοινωνιών, όπου έχει καταγράψει χίλιες περιπτώσεις ρωσικών παρεμβάσεων. Είναι λοιπόν μια πρόκληση η οποία μας αφορά όλους και αυτό το διαπίστωσε και η Κομισιόν. Η Task Force αυτή διευρύνεται, αλλά αρκεί. Λοιπόν, με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώς το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να μιλάμε λιγότερο και να κάνουμε περισσότερα. Και πρέπει η Κομισιόν να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μιλάμε για δύο συγκεκριμένα πράγματα μέσα, περισσότερα κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, περισσότερα λεφτά για αναλύσεις και έρευνα, περισσότερα λεφτά για εκστρατείες αντιπαραπληροφόρησης, για να μπορέσουμε να αμυνθούμε όλοι μας. Δεύτερον, οι γίγαντες της τεχνολογίας. Όταν μιλάμε για πλατφόρμες ε, όπως ε, το Facebook, είναι ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν, να υπάρξουν δεσμευτικοί κανόνες, όχι γενικοί κώδικες συμπεριφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράες για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Λίναρς μόλις είπε ότι είχαμε ένα ψήφισμα, μια συζήτηση και τώρα ξαναρχόμαστε και συζητάμε τα ίδια. Υπάρχει λόγος όμως γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι κάτι συμβαίνει δεν είναι κάτι το οποίο εμείς υπερβάλλουμε, όπου εμείς υπερβάλλουμε. Η Επίτροπος, η κυρία Γιούροβα και ο κύριος Κίνγκ δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και μήνες. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο και εμείς εργαζόμαστε, θέλουμε μια ειδική επιτροπή για κάποιο λόγο. Ο λόγος δεν είναι ότι ο Ντόναλτ Τραμπ ε, λέει στον Μπόρις Τζόνσον ε, ε, θέλω να αγοράσω το Εθνικό Σύστημα Υγείας σου ε, δεν μιλάμε για τέτοιου είδου ε, ε, παρεμβολέ. Αυτέ οι παρεμβολέ δεν μα αρέσουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όλο και πιο πολλά αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει παράνομη παρέμβαση, κρυφή παρέμβαση. Το είχε πει και ο Τζον Φιζαλ Κέναντι. Ένα να ψηφίσει διαφορετικά ε, τη δημοκρατία. Και αυτό φάνηκε και με την Cambridge Analytica. Αυτό είναι αντισυνταγματικό είναι κατά της νομολογίας σας. Είμαστε λοιπόν σαφείς γιατί πράγμα μιλάμε τελικά. Είναι κάτι παράνομο και είναι κάτι που γίνεται κρυφά. Αυτό σας πλήττει σήμερα, μας πλήττει σήμερα εμάς, αύριο θα πλήξει εσάς. Χαίρομαι που οι Βρετανοί συνάδελφοι ε, ξεκίνησαν τη συζήτηση αυτή, διότι εδώ ε, αποκαλύπτουμε τα τελευταία στοιχεία για το θέμα αυτό στη δική μου χώρα, από μια συντηρητική κυβέρνηση, ε, καλύπτει στοιχεία από το κοινό, δεν θέλει να αποκαλύψει τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τι διάφορε εκθέσει τη υπηρεσία ασφαλεία σε ό,τι αφορά τη ρωσική παρέμβαση. Και αυτό συμβαίνει και σε μεγάλε χώρε τη Ένωση. Είναι κάτι που έχει εγκριθεί από τι υπηρεσίε πληροφοριών ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να μην δημοσιευθεί. Παρ' όλα αυτά δεν δημοσιεύεται. Πόσα περαιτέρω στοιχεία χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι υπαρκτά. Ε, η Κομισιόν βεβαίω μιλάει για συνεχή ε, παραπληροφόρηση στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου, όπως και στις ΗΠΑ, όπως και στη Γαλλία. Η έκθεση αυτή μυρίζει, μιλάει για περιορισμένη δράση. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του νέου ρόλου της, με τη νέα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει όσα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα. Θέλουμε να υπάρχουν κλήσεις ασφαλείας online και offline. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με, τα, με τις ψευδείς λογαριασμούς, με τα στοιχεία προέρχονται από bots. Ε, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από, ε, από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι παράνομο, το οποίο γίνεται κρυφά και πρέπει να κάνουμε κάτι οπωσδήποτε για να προσπίσουμε τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφο Χόρουντ έχει το λόγο. Ναι, συγχαρητήρια για την εκλογή σας κυρία Αντιπρόεδρε και συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ για την ε, εισαγωγή σας αλλά από ό,τι κατάλαβα υποσχεθήκατε μια συντονισμένη απάντηση απέναντι στις ξένες παρεμβολές ε, πρέπει να είναι συντονισμένες ε, με τα κράτη-μέλη. Ε, είτε έχουμε Brexit είτε όχι. Ξέρουμε ότι επενδύονται ρωσικά χρήματα στον Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα και στο Λονδίνο και αυτό θα έπρεπε να μας δώσει μέσα πίεσης για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχουν ακόμα στοιχεία από τις υπηρεσίες ασφαλείας που δεν έχουν ε, δημοσιευθεί. Αναφέρθηκε ήδη αυτό. Αυτό δείχνει ότι η απάντησή μας δεν ήταν η κατάλληλη. Η ρωσική επιρροή ε, υπήρξε στο δημοψήφισμα. Ε, όπως είπε ο κ. Μωράες, ε, όμως το Εθνικό Κοινοβούλιο, ε, η κυβέρνηση προσπάθησε να το φημώσει, αλλά παρόλα αυτά δεν δημοσιεύει τη συγκεκριμένη έκθεση. Κανεί δεν είναι κατά τη έκθεση αυτή, τη έκθεση αυτή, μόνο ο Πρωθυπουργό. Και αυτό διότι ενδεχομένω η έκθεση αυτή να αναφέρεται στι δωρεέ ε, από Ρώσου προ το κόμμα ε, του κυρίου Τζόνσον και προς το, ε, στην καμπάνια υπέρ του Brexit. Ε, λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα έχει δώσει το Δημοκρατικό Φόρουμ, όπου μπορούμε να κρούσουμε τον κόσμο του κινδύνου και ελπίζω η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο αποφασιστική Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κούνκε έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ψηφιακές επιθέσεις είναι επιθέσεις ε, σχεδόν ε, ανύπαρκτες, γιατί μιλάμε για ένα εχθρό ο οποίος, εφευρίσκουν ένα εχθρό ο οποίος ε, δεν υπάρχει, αλλά αποτελούν μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή για τις δημοκρατικές αρχές επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αξίες μας. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να δράσουμε η Κομισιόν ε, είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο για αντιμετώπιση της ε, παραπληροφόρησης. Σας ευχαριστώ και είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνει πολύ πολύ περισσότερα. Το κομμάτι της ε, Europol, το οποίο ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, θα πρέπει ακριβώς να δει το τι γίνεται. Ε, κάποια μέτρα αρκούν, αλλά είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν αρκούν. Κάθε κράτος μέρος πρέπει να πάρει πολύ στα σοβαρά την απειλή των ε, ψηφιακών επιθέσεων, γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς εμάς πολιτικούς ε, σχετίζεται και με την προστασία από τέτοιες άπειλες. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να έχουν τις δυνατότητες για να λάβουν τις ε, ευθύνε τους και οι μεγάλες ψηφιακές ε, πλατφόρμες ε, να εργαστούν κατά των δυνάμεων αυτών που απειλούν την δημοκρατία μας. Σας ευχαριστώ. Χουχτασάρη για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η παρέμβαση στις ευρωπαϊκές εκλογές φυσικά θα πρέπει να αποτραπεί. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ο κόσμος να μπορεί να διακρίνει την ε, γνήσια ενημέρωση από την προπαγάνδα. Ε, είναι απαράδεκτο η Ρωσία, η Κίνα ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα να προσπαθεί να παρέμβει σε εκλογικές διαδικασίες υποσκάπτοντας ε, την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε τέτοια κατάχρηση. Και φυσικά ε, μερικές φορές ε, ο κόσμος αναζητά μια εναλλακτική λύση από τα παραδοσιακά κόμματα. Ο Ισλαμισμός, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια θέσεων απασχόλησης στη βιομηχανία, η υπονόμευση του κράτους ε, πρόνοιας, είναι λόγια τους οποίους ε, τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν τη δύναμη τους εκλογές. Οι πυροβολισμοί και βόμβες μερικές φορές ε, έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σκανδιναβικές χώρες. Γι' αυτό και τα εθνικιστικά κόμματα κερδίζουν έδαφος, γιατί θέλουν να ανακτήσει την ασφάλεια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ πιστεύω σε μια καλύτερη και ασφαλέστερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συγχαρητήρια για την επανακλογή σας. Θα έχετε πολλά να κάνετε στα νέα σας καθήκοντα. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες χρήσης διπλών μέτρων και σταθμών. Πολλοί συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο μίλησαν ε, για παρεμβολή από ξένες δυνάμεις. Αυτό όμως όταν δεν σας ενοχλεί το εντοπίζετε όπως γίνεται με τους stories στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν όμως χρηματοδοτούνται κάποιες καμπάνιες από το δισεκατομμυρίουχο όρος, τότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιείτε διπλά μέτρα και σταθμά. Ή θα είστε κατά της ξένης παρέμβασης, είτε θα την αποδεχτείτε. Αλλά όταν εντοπίζετε ξένη παρέμβαση θα πρέπει να τη στυλιτεύετε από όπου και αν προέρχεται. Σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Γι' αυτό έγραψε ο Τζόρτζ Όργουελ για το Υπουργείο της Λογοκρισίας, Υπουργείο της Αλήθεια. Για σας έγραφε όταν έγραφε τα βιβλία του Τζόρτζ Όργουελ, γιατί πραγματικά είστε ε, οι πρωταθλητέ των διπλών μέτρων και σταθμών. κυρία Περέρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η προάσπιση της δημοκρατίας ε, απαιτεί πολύμορφα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση και την ανεξαρτησία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέναντι στο συγκεντρωτικό μονοπόλιο ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών της ενημέρωσης ε, και ο σεβασμός των διοντολογικών και ηθικών αρχών και κριτηρίων. Και μάλιστα η συγκέντρωση που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κυρίαρχων πολιτικών και των μεγάλων πολυεθνικών. Ε, ουσιαστικά όμως έτσι περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης ε, και εξαπλώνονται και διαδίδονται ε, ψευδείς ειδήσει ε, και μόνο ιδέες που σας εξυπηρετούν. Ουσιαστικά έτσι ενισχύεται ο λαϊκισμός και ο σκοταδισμός και ανοίγουν οι πόρτες προς τις ακροδεξίες απόψεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μερικές φορές χρησιμοποιούμε προσχήματα για να συγκαλύψουμε αυτή την πραγματικότητα και ακολουθούμε ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο της ενίας και αντιδραστικής σκέψης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κυρία Αντιπρόεδρε. Δικαίως η Ούρσουλα Φαντερ σήμερα ανέφερε τους πολλούς Τσέχους και Σλοβάκους που πριν από 30 χρόνια πάλεψαν για την ελευθερία στην Πελούδινη Επανάσταση και χάρη σε αυτήν την μάχη η ελευθερία και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι κάτι το οποίο πλέον υπάρχει σε όλη την Ευρώπη αλλά είναι και κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε και πρέπει να αναλάβουμε δράση, γιατί απειλούμαστε. Το θέμα δεν είναι μόνο μια συζήτηση για τα ψέματα του Brexit, είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Και το βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε ευρωεκλογέ και σε εθνικές εκλογές. Μάλιστα, το κοινοβούλιο αυτό ενέκρινε ένα ψήφισμα τον προηγούμενο μήνα για το πώς θα προσεγγίσει καλύτερα την καταπολέμηση των ξένων παρεμβάσεων και της παραπληροφόρησης είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για πολιτική δράση. Θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα που θα περιμέναμε από την Κομισιόν. Πρώτον, η καταπολέμηση των ξένων παρεμβάσεων και της ε, παραπληροφόρησης πρέπει να γίνει πολιτική προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της ε, Κομισιόν τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να γίνει πολιτικό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο να μιλάμε για το ποιο ε, φταίει και ποιος, ε, ποιον πρέπει να κατηγορήσουμε. Και πρέπει να υπάρξει κάποια αρρύθμιση. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ασφαλές διαδίκτυο, τι αξίε της Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημοκρατία μα και να ρίξουμε περισσότερα χρήματα στην εκπαίδευση ε, ειδικά στον τομέα που είναι πιο ευπαθής οι πολίτες μας ε, στο διαδίκτυο, στον ψηφιακό χώρο και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μποναφέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη όντω έχει εγκρίνει ένα ψήφισμα τον Οκτώβριο μετά την πρωτοβουλία της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για να καταδικάσουμε τις παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά εντωμεταξύ η Ιταλική δικαιοσύνη προσφάτως ξεκίνησε μία έρευνα για διεθνή διαφθορά για την ρωσική χρηματοδότηση της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνη. Αλλά πέρα από αυτό ε, υπάρχουν ε, και στοιχεία τα οποία ποτέ δεν έχουν ξεκαθαριστεί εις βάθος. Είχε προηγηθεί η περίπτωση της Αυστρίας, η περίπτωση της Γαλλίας και πιο πρόσφατα είχαμε και παρεμβάσεις ε, βεβαίως στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά δεν είναι συνωμοσιολογία, είναι πραγματικά επικίνδυνα για το δημοκρατικό μας σύστημα, γιατί συχνά βλέπουμε κάποιες εκστρατείες μη στο διαδίκτυο τα οποία επηρεάζουν την κοινή γνώμη και άρα την εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό η συζήτηση αυτή να συνεχιστεί. Θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι έχουμε το καθήκον να υπερασπιστούμε τα δημοκρατικά μας θεσμικά όργανα και να είμαστε ξεκάθαροι. Σα ευχαριστώ. Λουαζό για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού μοντέλου είναι να επιλέγουμε ποιου μα κυβερνούν. Όμω όλο και πιο συχνά βλέπουμε ξένε δυνάμει που προσπαθούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών μα. Ο στόχο είναι προφανή, να αποδυναμωθούμε. Το διαπιστώνουμε αυτό, λυπούμαστε γι' αυτό, το καταδικάζουμε, αλλά μιλάμε πραγματικά για έναν καρκίνο, ο οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να καταστρέψει τον ελεύθερο κόσμο μα. Πρέπει όμω να δράσουμε και να δράσουμε γρήγορα. Γιατί να μην δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας των δημοκρατιών έτσι ώστε κάθε κράτο μέλο να μπορεί να λάβει την απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσει τι κυβερνοεπιθέσει, τι χειραγωγήσει και την παραπληροφόρηση που ε, έχουν ως στόχο τις εκλογικές διαδικασίες. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, ε, Προστασίας Διατροφικής Διατροφική ασφάλεια. Εάν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά που βρίσκονται στο πιάτο μα, πρέπει να μπορούμε να προστατεύσουμε και αυτά που περνάνε από ε, τις κάλπες μας και από τις ψήφου μα, τα ψηφοδέλτιά μας. Ε, οι επιπτώσει είναι εξίσου σοβαρέ ε, από τη, τη δηλητηρίαση, την πολιτική, από ότι από την ε, διατροφική. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σας συγχαίρω μάλλον για την εκλογή σας κυρία Αντιπρόεδρε και χαίρομαι που δεσμεύεστε για να προστατεύσετε τις δημοκρατίες μας. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Άλλαρ για δύο λεπτά. Thank you Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, και εγώ να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Εγκρίναμε το ψήφισμα τον Οκτώβριο και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ξανασυζητάμε, διότι πολλά πρέπει να γίνουν. Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι αποδεκτό ότι η ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016 έλαβε χώρα. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό. Ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Τζόνσον, την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ποτέ δεν, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ρωσία παρενέβη στις δημοκρατικές ε, εκλογικές διαδικασίες ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017 όμως ε, ο Υπουργό Εξωτερικών του ΕΒ, ο κ. Τζόνσον τότε, είπε ότι είχε δύο αποδεικτικά στοιχεία ρωσική παρέμβαση ε, στι δημοκρατικέ διαδικασίε ε, του ΕΒ. Βασιλείου. Τελικά, ποιο Μπόρι Τζόνσον λέει την αλήθεια. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό τη Σκωτία σήμερα, είναι επικίνδυνο ο κ. Τζόνσον και δεν είναι κατάλληλο, είναι ακατάλληλο για την ε, Πρωθυπουργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κλίμα ξενοφοβία, ρατσισμού απέναντι στου ξένου και χαίρομαι για αυτά που ακούω σήμερα. Διότι με το κείμενο που ψηφίσαμε νωρίτερα φέτος θα πρέπει πλέον να μπορούμε να επανέλθουμε στην υπόθεση αυτή και να προσέχουμε τι λόγια χρησιμοποιούμε. Βεβαίως υπάρχουν ε, κρατικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την παρέμβαση. Εγώ ω Γάλλο πολίτη που εκπροσωπεί τη Σκοτία σε αυτό το κοινοβούλιο, πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε την παρέμβαση των ξένων κρατών. Ας, θα πρέπει να ανοίξουμε τη δημοκρατία μα για όλου του πολίτε που ζουν εδώ, μεταξύ των οποίων και ξένοι όπω εγώ. Ε, Στι μελλοντικέ εκλογέ δεν θα μπορέσω να ψηφίσω για το Westminster, αλλά εύχομαι σε όλου του συναδέλφου καλή τύχη, ιδιαίτερα του ευρωβουλευτέ εδώ και, και όλο ιδιαίτερω ε, τον συνάδελφο Άλαν Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ακούγεται πολύ φασαρία εδώ. Ξέρετε, η ακουστική στο κτίριο αυτό είναι απίστευτη, οπότε όπου και να μιλάτε, ακούγεστε. Προσπαθήστε λοιπόν να μιλάτε χαμηλόφωνα, ακόμα και στο γείτονά σας. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τέρτς. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, λάθος σας. Ο κύριος Μαριανή έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ε, μην με ξεχνάτε πρόεδρε. Στη Γαλλία μετά το 1870 υπήρξε ένας τρόμος ε, για τους βουλευτές, για τα, στις εφημερίδες. Λέγαμε ότι η Γερμανία επηρέαζε τις εκλογές μας. Υπήρχε ένα άλλο το χέρι τη Γερμανία. Ορισμένε φορέ αυτή η φόβη είναι βάσιμη, αλλά συχνά πρόκειται απλά για φαντασιώσει. Είναι η αίσθηση μια ανάγκη εθνική ενότητα για να υπερασπίσουμε τι πατρίδε μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά είναι, έχει μια παράδοξη στάση αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρεί ότι κάθε επιστροφή στην εθνική συνείδηση είναι επικίνδυνη και ταυτόχρονα θέλει να μα προστατεύσει από τι ξένε επεμβάσει. Οποιαδήποτε συζήτηση για παρέμβαση ξένων δυνάμεων στι εκλογέ στην πραγματικότητα είναι σαφή, μια σαφή πολιτική επίθεση απέναντι στα πατριωτικά κινήματα τα ευρωπαϊκά και απέναντι στη Ρωσία που θεωρείται ότι παρεμβαίνει ε, στις εκλογές μας και παραπληροφορεί στις δημοκρατικές διαδικασίες ε, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές. Υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις άμεσης παρέμβασης, σαφής, σαφούς παρέμβασης από ηθήνοντες ή από οι ομάδες πίεσης σε πρόσφατες εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σόρος και η Open Society ε, στους στίχους της Βουδαπέστης κάνει προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης. Στην Αλγερία ζητείται ε, να, να καταργηθεί ε, το κόμμα μας. Ε, στη Γερμανία δίνονται οδηγίες για το που θα ψηφίζουν άτομα που έχουν διπλή υπηκότητα. Η υποστήριξη των κύριο Μακρόν δύο μέρες πριν τις εκλογές από τον κύριο Ομπάμα. Βγαίνουν από μια συνεδρίαση όπου ζητείται μεγαλύτερη υποστήριξη στην αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Πριν κατηγορήσουμε τους άλλους να δούμε και τι κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέρμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια στην Επίτροπο Γιώροβα για την επανεκλογή της. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις παρεμβάσεις. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις. Είχαμε και στην Καταλωνία από Ρώσους πράκτορες. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες παρεμβολές. Αλλά παρεμβάσεις είχαμε πολύ άριθμες και στην Ευρώπη. Είχαμε τι παρεμβάσει της κυρίας Μέρκελ, για παράδειγμα, σχεδόν σε όλες τις ε, εκλογές, ε, τι ευρωεκλογέ ε, που έγιναν στην Ευρώπη. Μαζικά, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία, είχαμε τέτοιε παρεμβάσεις. τι παρεμβολές, τι παρεμβάσεις έγιναν από τις Ευρωπαίους προ προς τις Ηνωμένε Πολιτείες ο, στις πρόσφατες εκλογές όταν όλοι σαν χοροδία προσέβαλαν τον Τραμπ. στην Ισπανία αυτή τη στιγμή το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα δημιουργήσει ε, εκλογικό συνασπισμό με, τη, με τους κομμουνιστές του Ποδέμος που είναι ουσιαστικά ε, ένα franchise το Ποδέμος από τη Βενεζουέλα. Το χρηματοδότησαν και το σχημάτισαν ε, οι Βενεζολάνοι του Τσάβες με τους Κουβανούς. Και ουσιαστικά θα έχουμε το Μαδούρο στο Συμβούλιο Υπουργών μας στην Ισπανία. Και αυτό γίνεται με την ανοχή των αποσχεστών. Και μάλιστα είχαμε αυτή τη μαζική παρεμβολή που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Λατινική Αμερική. Τώρα θα έχουμε αντίστοιχα από τη Λατινική Αμερική μέσω των κομμουνιστών παρεμβολή στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα, στην συνάδελφε, να σας δώσω το λόγο για δύο λεπτά. Δεν τα έχω τα γερμανικά. Δεν τα έχω περάσει. Δεν, τα έχω περάσει. Λοιπόν, το θέμα της παρέμβασης κατά της ανεξαρτησίας είναι ένα πρόβλημα, αλλά λέγονται και διάφορα ψέματα. Τα εξετάζουμε όλα αυτά. Η διάδοση λοιπόν της παραπληροφόρησης είναι μια διάδοση ψευδών. Κανείς από εμά δεν είναι κατά των ελευθερών μέσων ενημέρωση. Κανείς δεν ε, αντίσταται, αλλά όλοι μας ε, γνωρίζουμε ότι στα κοινωνικά δίκτυα διαδίδονται ψέματα και λάθος πληροφορίες ε, και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τσεχική δημοκρατία είχαμε παρακολούθηση από, την ε, μυστική, από τις μυστικές υπηρεσίες ε, της Κίνας και της Ρωσίας ε, και διαβάζουμε ότι υπάρχει και μια προκλογική εκστρατεία με στόχο να αποδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιρροή των πολιτικών διεργασιών στόχος είναι να διχάσουν μεταξύ τους τα ευρωπαϊκά κράτη και στη Μεγάλη Βρετανία τα κατάφεραν. Άρα δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει είναι να παρεμποδίσουμε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων επενδύσεων. Εμείς ε, θέλουμε έχουμε ε, ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Προφανώ και το θέλουμε αυτό. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίζουν τα δημόσια μέσα ενημέρωση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να καλούνται να εφαρμόσουν μια οδηγία ε, για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση για τα δικαιώματα των δημιουργών. Άρα δηλαδή πρέπει να στηρίζονται οι δημιουργοί και τα καλά μέσα ενημέρωση ήθελα να υποστηρίξουμε και καλύτερα την Stratcom. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει ε, συγκεκριμένες ε, δυνατότητες αντιμετώπισης της Κίνας και της ε, Ρωσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ρούις Ντεβέσα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από πλευράς μου στην κυρία Γιούροβα που ε, είναι πλέον νέα επίτροπος. Έχουμε θέματα πολλά επί των οποίων θα συνεργαστούμε μεταξύ άλλων των σημερινών. Γι' αυτό το σημερινό θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι, οι, πολιτικοί θύνοντες, θα πρέπει να παράψουμε να παρασταίνουμε τους ε, άσχετους γιατί υπάρχει σαφώς μία συμμαχία εχθρών εκτός της Ένωσης που προσπαθούν να την αποδυναμώσουν και ακόμα και να την καταστρέψουν και που μάλιστα συμμαχούν με ανθρώπους εντός των κρατών μελών μας και που σχηματίζουν κινήματα πολιτικά ή άλλες δομές. Και αυτό είναι πραγματικότητα και πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και να την εξαρθρώσουμε. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις ώστε ξένες δυνάμεις να χρηματοδοτούν προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωεκλογές. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τον ίδιο βαθμό προστασία στα κράτη-μέλη, γιατί και μέσα από τα κράτη-μέλη μπορούν να δράσουν. Ευχαριστώ πολύ και να βλάψουν την Ένωση. Ευχαριστώ. Νεσίγκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη για τον Αμένο Βασίλειο όπου το θέμα της παρεμβάσεως στις εκλογές είναι πραγματικά σε υψηλό σημείο στη, στο πρόγραμμα συζητήσεων. του Συντηρητικού Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταμόρφωσε τα τελευταία χρόνια, μεταμορφώθηκε πέραν αναγνωρίσεως τα τελευταία χρόνια και πολλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για επηρεασμό από τη Ρωσία και από τη ΣΥΠΑ για τη, τη μεγάλη αλλαγή. Οι δωρές από τους Ρώσους ολιγάρχες και τις γυναίκες τους ε, είναι πολύ σημαντικέ. 200.000 αυτή την εβδομάδα και μόνο την πρώτη τη προεκλογική εκστρατεία. Βαθιέ τσέπε που προσπαθούν να επηρεάσουν τι εκλογέ. Πάντα τα έκαναν, αλλά η κλίμακα και η τεχνολογία είναι κάτι πρωτοφανέ. Ο αντίκτυπο παραπληροφόρηση αναγνωρίστηκε από σοβαρού ερευνητέ που κατέδειξε ότι εκείνοι που έχουν τροφοδοτήσει, ε, έχουν μάθει αυτές οι ειδήσει, είναι δύσκολο να τους αλλάξει γνώμη και να τους ενημερώσει. Ε, αυτοί που το μαθαίνουν για πρώτη φορά. Λοιπόν, είχαμε ασφάλεια τα τελευταία χρόνια από τον ψυχρό πόλεμο και χαλαρώσαμε όσον αφορά τον κίνδυνο τη ξένη προπαγάνδα. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Είναι σοβαρέ οι απειλέ που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίε μα. Αυτό σημαίνει η δημοσίευση των ε, φακέλων της Ρωσίας στον Ηνωμένο Βασίλειο και να αναλάβουν την ευθύνη, την ευθύνη τους στα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να εξακριβώνουν να είναι αληθή αυτά που πρόκειται να τυπώσουν και να προβάλλουν. Ευχαριστώ. Κύριε Ρόουετ, για ένα μισή λεπτό. Κυρία Ρόουετ, μάλιστα. Ε, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κάποτε ε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο μαζί με την Αθήνα ήταν ε, τα δίδυμα αρχέτυπα για τη δημοκρατία αλλά κάθε δημοκρατία χρειάζεται μέτρα διαφύλαξης και θα πρέπει οι κυρώσει ε, να ε, επιβάλλονται στους αναδυόμενους ολιγάρχες. Αν διαφυλάξει ε, όταν τα μέλη στο Κοινοβουλίο ήταν κάποτε ε, δεν ήταν τσάκα δεξιά στο κοινοβούλιο παλιά στον Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα όμω έχουν περάσει οι κυρίε και βλέπουμε πώ οι οπαδοί του Μπόρι Τζόνσον δεν αφήνουν να δημοσιευθούν οι φάκελοι για τη Ρωσία. Ε, διαγράφονται τα ονόματα των εμπλεκομένων και δίνουν σε λόμπις, ε, παίρνουν ε, από, χρήματα από λόμπις για να μπορούν να παρέμβουν και δεν ε, δημοσιεύουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για παρέμβαση του κόμματος στις εκλογές του 2016. Όλα αυτά θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν πριν ξεκινήσουν οι νέες εκλογές που χαρακτηρίζονται από πάρα πολλά χρήματα που δίνονται, παραπληροφόρηση από τα ίδια άτομα που πραγματοποιούν αυτή την παραπληροφόρηση. Στην αρχαία Αθήνα ε, μπορούσαν να ε, ε, ο Δήμος μπορούσε να εξωστρακίσει όποιον απειλούσε το κράτος δικαίου στην αρχαία Αθήνα και τον εμπόδισαν να αναλάβει πολιτικά αξιώματα για μια δεκαετία. Η σύγχρονη δημοκρατία επίση θα έπρεπε να έχει ένα αξιοπρεπέ εργαλείο να κάνει αυτή τη δουλειά και θα πρέπει να συμπεριλαβεί και τον αποκλεισμό από την πολιτική, διότι για του πάρα πολλού πλούσιου του επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή δεν του αγγίζει καν συνάδελφε Αρντώνε, για 1,5 λεπτό. Πραγματικά, Πρόεδρε, μιλάμε για νιωστή φορά για τις παρεμβάσεις άλλων χωρών στη δική μας δημοκρατία και στις εκλογές μας. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό είναι ε, τραγικοκομικό, κομικοτραγικό φαινόμενο. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στο θέμα συμφορία του Brexit, μιλάμε για τον Μπολσονάρο, για τον Τραμπ και βλέπουμε ότι άμβοψε η λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και στις ευρωεκλογέ και διαρωτάστε ε, πώς είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά. Για σας είναι ένα μυστήριο. Λοιπόν, ψάξτε, ψάχνετε να δικαιολογήσετε τη λαϊκή ψήφο ε, ε παράλογες συνωμοσίας και ε, πηγαίνετε να ξυπνήσετε, διότι εμείς είμαστε η παραγωγή, θεωρείτε, των fake news. Κρίμα όπου εσείς δίνετε ψευδείς ειδήσει με την φιλοευρωπαϊκή σας προπαγάνδα που πληρώνετε από τους ε, φορολογούμενους.